συμμετέχοντα μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. ψηφοφορία αύριο στις 11.30. Και τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε την έκθεση της Edith Bauer για την κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης. Δίνω το λόγο λοιπόν στην εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όμως έχετε προσέξει ότι στις οθόνες δεν μπορούμε να δούμε γυναίκες εισηγήτριες άνω των 50 ετών. Μήπως έχετε προσέξει ότι είναι πολύ λιγότερες οι γυναίκες άνω των 50 από τους άνδρες. Οι στατιστικές καταδεικνύουν ότι παρά το γεγονός ότι 55% των ανδρών είναι ενεργοί στην αγορά εργασίας, το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόνο 40% για τις γυναίκες άνω των 50 ετών. Αν προσπαθήσετε να δείτε σχετικά στατιστικά στοιχεία, βρίσκεται στατιστικά στοιχεία μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Αυστραλία και είναι ελάχιστα τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα κοινοβούλια περνάει συνεχώς νομοθεσία για να αυξηθεί το όριο συνταξιοδότησης, αλλά παρόλα αυτά διαπιστώνεται ότι ο κόσμος αποχωρεί από την αγορά εργασίας νωρίτερα. Η στρατηγική του 2020 έχει στόχο να έχουμε ένα ποσοστό απασχόλησης 75% και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Επομένως, δικαίως μπορούμε να ρωτήσουμε τι θα πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ε, αποχωρεί νωρίτερα ο κόσμος από την αγορά εργασίας. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες αφήνουν την αγορά εργασίας. Πολλές φορές ε, βρίσκονται αντιμέτωπες με διάφορες διακρίσεις. Δεν πρόκειται μόνο για μία, πρόκειται για ένα περίπλοκο σύνολο ε, διακρίσεων και μία εκ των διατρήσεων είναι η γύρανση. Γι' αυτό δεν βλέπουμε γυναίκες σε τηλεοπτικές οθόνες άνω των 50 ετών και δεν πρόκειται για το μόνο τομέα στον οποίο έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα. Υπάρχουν επίσης και κοινωνικοί λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες αφήνουν την αγορά εργασίας. Μπορεί να πρέπει να φροντίσουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους αλλά μπορεί να οφείλεται και σε λόγου υγεία. Γι' αυτό λοιπόν και θα μπορούσαμε να έχουμε προληπτικά μέτρα για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Μία εκ των πολύ ασθενειών, για παράδειγμα, είναι η στεοπόρεση. Η κίνδυνη στον τομέα της εργασίας επίσης είναι ένας ε, από τους λόγους. Το 2012 είναι το έτος ενεργούς ε, γύρανσης και θα μπορούσαμε να έχουμε πρωτοβουλίες ε, προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν πολύ σεβαρός ε, συνέπειες διότι στην ηλικία των 50 ετών αυξάνεται το χάσμα μεταξύ των μισθών ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν ε, πολλές ε, επικίνδυνες ε, εργασίες για τις γυναίκες, επισφαλής εργασία επίσης και αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες ζουν σε κατάσταση μεγαλύτερης φτώχειας σε σχέση με τους άνδρες αντίστοιχης ηλικίας. Υπάρχουν βεβαίως οι διακρίσεις που είναι ένα γνωστό πρόβλημα αλλά σε μια έρευνα που έγινε ε, οι γυναίκες ε, στην πλειονότητά τους απάντησαν ότι οι διακρίσεις είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Επίσης υπήρχαν ε, και συμπεράσματα τα οποία καταδεικνύουν ότι η πρόληψη είναι φθηνότερη από την θεραπεία για τα συγκεκριμένα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξει μια λευκή βίβλος η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των γυναικών. Δεν μπορεί οι γυναίκες να μένουν ανασφάλιστες, για παράδειγμα, κατά τις περιόδους στις οποίες φροντίζουν τα παιδιά τους ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι οι οποίοι επιδεινώνονται με την ηλικία ε, και βάσει και των δημογραφικών τάσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και αν δεν γίνει κάτι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει στον τομέα της απασχόλησης και της καταπολέμησης της ένδυας για τη στρατηγική του 2020. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κλάς. Er ε, στην έκθεσή της η Έντιτ Bauer είναι πολύ συγκεκριμένη. Η κατάσταση των ηλικιωμένων γυναικών ε, χειροτερεύει δραματικά. Ε, ε, επιδεινώνονται στα προβλήματά τους όταν είναι χαμηλόμιστοι και οι γυναίκες. Ε, οι αποδοχές είναι μικρότερες, η ανεργία είναι υψηλότερη στις γυναίκες από τους άνδρες. Ε, τέσσερις φορές περισσότερο έχουν μερική απασχόληση, εργάζονται αλλά δεν πληρώνονται πάντα. Το χαμηλό εισόδημα των γυναικών έχει αντίκτυπο και στην σύνταξη που οδηγεί στην φτώχεια. Η έκθεση εξετάζει τα θετικά σημεία ε, το, ε, ο βαθμός που πλουτίζουν οι ηλικιωμένοι μια κοινωνία. Πολλές φορές παραβλέπεται αυτό και δεν γίνονται οι προσπάθειες που πρέπει. Οι κοινωνικές προκλήσεις σήμερα είναι να βοηθήσουμε να είναι ε, αξιοπρεπείς στη ζωή τους οι άνθρωποι αυτοί και ε, ακόμα και μετά τη συνταξιοδότηση θα πρέπει να μένουν υγιείς, δραστήριοι ε, και ε, ανεξάρτητοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μικολάζικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται από το εργατικό της δυναμικό. Η παράταση της, ε, του χρόνου εργασίας θα πρέπει όμως να είναι ορθολογική, ούτως ώστε οι συνθήκες εργασίας ε, να παραμείνουν ε, αξιοπρεπείς για τον άνθρωπο. Τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες, οι κοινότητες θα πρέπει να στηρίξουν τις γυναίκες ως επιχειρηματίες, να στηρίξουν παράλληλα και την ενεργό γύρανση και θα πρέπει μεταξύ των δύο προγραμμάτων να δημιουργηθούν συνέργειες. Έτσι θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, στις γυναίκες ε, που παρέχουν φροντίδα και πληρώνονται ελάχιστα ενώ φροντίζουν ε, δύσκολα περιστατικά. Ε, θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Ευχαριστώ κυρία Ντανσίλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η αλληλεγγύη μεταξύ γενεών και η χρήση του δυναμικού των ηλικιωμένων γυναικών είναι υψή τη σημασία. Πρόκειται για ένα πολύτιμο πόρο και ένα απόθεμα εμπειρίας που θα μπορούσε κάλλιστα να υποστηρίξει την όλη κοινότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στη βελτίωση των ίσων ευκαιριών και των πολιτικών που θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε τις διακρίσεις και τις ε, διακριτικές συμπεριφορές προς τις γυναίκες που πλησιάζουν το ηλικία συνταξιοδότησης. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την επιστροφή στο χώρο εργασίας μετά τη γέννα και τη δυνατότητα ε, να αλλάξει κάποιος τη θέση εργασίας τους ώστε να μην υπάρχουν κενά ε, εργασίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιγκερέιδο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων γυναικών είναι από τα μεγαλύτερα κοινωνικά μας προβλήματα και ένα μεγάλο αίτιο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Πολύ συχνά οι γυναίκες αυτές είναι τα θύματα χαμηλών αποδοχών, ανεργίας, προσωρινής και επισφαλούς εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιβιώσουν σε καταστάσεις μεγάλης κοινωνικής ευαλωτότητας και φτώχειας. Σε μια εποχή όπως η σημερινή, η κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση πρέπει να μας απασχολήσει για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ε, πέσουν θύματα διακρίσεων επειδή έκαναν παιδιά ε, σε μια ηλικία όπου δεν μπόρεσαν να γίνουν ανταγωνιστικές στο επάγγελμα ε, όπως θα μπορούσαν. Θα πρέπει η συνταξιοδότηση να γίνει με τρόπο αξιοπρεπή χωρίς διακριτική βία σε βάρος τους. Χρειάζεται υψηλή ποιότητα δημοσίων υπηρεσιών εδώ και ευαίσθητη χειρισμή σε τομείς όπως η υγεία και η στέγη. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση και που πρέπει να τα προσέξει ιδιαίτερα η Κομισιόν. Κυρία Φλαζίκοβα, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η παρούσα έκθεση ασχολείται με τις γυναίκες πριν από την συνταξιοδότηση, ηλικίες δηλαδή 55 με 64. Τα δεδομένα δείχνουν ότι στις 21 χώρες, σε χώρες μέλη το ποσοστό ε, αποδοχών είναι 20% χαμηλότερο από ό,τι των ανδρών. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη ισορροπίας σε βάρος των γυναικών πριν από την ε, συνταξιοδότηση. Αυτό ε, ανάγεται σε πολλούς κοινωνικούς παράγοντες. Οι διακρίσεις σε βάρος αυτών των γυναικών πρέπει να σταματήσουν. Αυτό αποτελεί, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των κρατών μελών, ούτω ώστε να ε, ενισχυθεί ο ρόλος του στην αγορά. Απευθυνέται στην Κομισιόν για να θεσπίσει κανόνες για τα κράτη-μέλη που θα βοηθήσουν τις γυναίκες ε, να ε, παραμείνουν δραστήριες στην αγορά εργασίας ε, και να έχουν και αξιοπρεπείς συντάξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νεβιτάλοβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα τομέα όπου έχουν, γίνονται διακρίσει ε, είναι η αγορά εργασίας. Δεν έχουν δικαίωμα ισότιμο στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε πολλέ άνεργε και νέες και ηλικιωμένες. Ε, αυτές οι δύο κατηγορίες υφίστανται τις περισσότερες διακρίσεις γιατί αναγκάζονται σε μερική απασχόληση. Μην ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα οι ηλικιωμένες γυναίκες συμβάλλουν πάρα πολύ στην ε, κοινωνία, στην κοινωνική ζωή. Πολύ συχνά ε, εργάζονται χωρίς αμοιβή, φροντίζουν παιδιά και εγγόνια και οι γυναίκες αυτές εργάστηκαν όλη τη ζωή τους και όταν είναι, είναι ηλικιωμένες και υγιείς θα πρέπει να εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα να εργαστούν. Καλό λοιπόν την Κομισιόν και του χρόνου, το χρόνο, το έτος της ενεργού γύρανσης, να λάβει μέτρα για να βοηθήσει τις γυναίκες αυτές, ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας. Ευχαριστώ κύριος Μεστσάρος. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ήθελα να λάω το λόγο, αλλά αν επιμένετε κάτι μπορώ να πω. Η κυρία Παπαδοπούλου. Το μικρόφωνο σα. Μάικρο. Κυρία Πρόεδρε, είναι γεγονό πω τα ηλικιωμένα άτομα ηλικία 55 με 64 ετών υφίστανται τον ηλικιακό ρατσισμό, ηλικιακέ διακρίσει. Οι γυναίκε ιδιαίτερα βιώνουν αυτέ τι διακρίσει, αλλά έχουν επιπρόσθετα και τις άλλες εύφυλες ε, διακρίσεις λόγω φύλου, στερεότυπων αντιλήψεων, επισφαλούς υγείας ή αναπηρίας. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι το 2012 θα είναι έτος ενεργού στήριξης γιατί δίνει μια μοναδική ευκαιρία περαιτέρω ευαισθητοποίησης για την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της ηλικίας σε όλες τις πολιτικές για να αποφευχθεί ακριβώς ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο κάθε λογής ρατσισμό ενάντια στα άτομα τριτή ηλικία. Σε μια Ευρώπη που γερνά δεν έχουμε την πολυτέλεια να θεωρούμε τη γύραση του πληθυσμού ω κοινωνικό-οικονομικό βάρος. Αντίθετα έχουμε υποχρέωση να καταπολεμήσουμε τι προκαταλήψει, να στηρίξουμε την ενεργό με προγράμματα και δραστηριότητε και να διασφαλίσουμε την ίση πρόσβαση όλων στη υγειονομική περίθαλψη και στη μακροχρόνια φροντίδα. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Ταγιάννη, παρακαλώ. Θα ευχαριστήσω πρώτα την κυρία Μπάουερ για την εκπόνηση της εκθέσεως. Η οικονομική ανεξαρτησία για άνδρες και γυναίκες είναι στόχος μας για το 2015 για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Στόχος μας είναι η αύξηση της απασχόλησης για άνδρες και γυναίκες και εθνικών πολιτικών δηλαδή που έχουν ως στόχο να αυξήσουν την απασχόληση των γυναικών και να μειώσουν τις ε, ανισότητες μεταξύ άνδρων και γυναικών και ιδίως άνω των 50 ετών. Οι γυναίκες οι οποίες πλησιάζουν το συνταξιδοτικό όριο ηλικίας βρίσκονται σε ιδιαίτερη κατάσταση διότι είναι ενίδικα τα παιδιά αλλά στις οικογένειες συχνά φροντίζουν τους ηλικιωμένους γονείς. Η επαγγελματική τους και η ιδιωτική τους ζωή είναι απαραίτητο να μπορεί να συγκεραστεί, διότι αλλιώς οι γυναίκες αυτές χάνουν πολλά δικαιώματα. Η... Κάνει λοιπόν σημαντική προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόθεση των στόχων αυτών και με τη γονική άδεια και την άδεια πατρός δηλαδή και ούτω καθεξής. Έχουμε αναθέσει μελέτες για να ελεγχθούν τα αποτελέσματα των ε, διαφόρων αυτών τύπων αδειών και τα αποτελέσματα τα αναμένουν περί το τέλος του έτους. Μετά από αυτό θα μελετήσει τα μέτρα που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, οι γυναίκες άνω των 75 ετών βρίσκονται σε σημαντική και ε, σε σημαντικά επικίνδυνη θέση από άποψη υγεία περισσότερο από τους άνδρες και συχνά έχουν ανεπαρκή συντάξει. Συχνά επίσης αυτό οφείλεται και στην βραχύτητα της επαγγελματική του σταδιοδρομίας. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να διορθωθεί. Η θέσπιση ίδιου ορίου ηλικίας συνταξιδοτήσεως και για άνδρες και γυναίκες είναι ένα μέσον για να καταλήξουμε στο στόχο αυτό έτσι επίσης ώστε να διασφαλίζεται η απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, για παράδειγμα και στη διάρκεια της ε, ε, μητρότητας με στόχο να βελτιωθούν οι διατάξεις για τη συντάξη των γυναικών. Του χρόνου θα εξετάσουμε μαζί με τις ε, χώρες μέλη τη ρύθμιση των ε, συνταξιοδοτικών συστημάτων και θα υποβάλουμε και έκθεση για την γύρανση με ιδιαίτερη, ιδιαίτερο στόχο τις γυναίκες που βρίσκονται σε ηλικία συνταξιδότησης με χαμηλό ίσμα. Τους επόμενους μήνες θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά, να συνεργαζόμαστε μάλλον στενά με τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναμένουμε την δική σας δέσμευση που θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε μέτρα με για την καλύτερη δυνατή συμβολή έτσι ώστε να είναι ενεργός η γύρανση για να αντιμετωπίζονται οι δημογραφικές ε, αλλαγές. Αφόσον τώρα ε, θα μπουν στην τρίτη ηλικία τα μέλη του περίφημου Baby Boom. Αυτά θα είναι μια σημαντική ε, ευκαιρία για να συζητήσουμε θέματα γυράσκοντος πληθυσμού και να καταδείξουμε τον πλούτο που μπορούν να προσφέρουν οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, της ε, ηλικιακής αυτής ομάδας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση, η ψηφοφορία αύριο στις 11.30. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί, 3η 13 Σεπτεμβρίου του 2011, στις